Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης είναι πλέον διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι. Επομένως εγκρίνονται τα πρακτικά. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε κοινή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με πρώτη έκθεση την έκθεση της κυρίας Φερέιρα. Να δώσουμε το λόγο λοιπόν all'onorevole Schwab. Στον Schwab. Prego. Εκπλήσω με πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο.